Καλησπέρα σε όλους. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα χτεσινά πρακτικά στη διάθεσή μας. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Πρώτη συζήτηση για το απόγευμα είναι